Αδελφοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας για την κατάσταση στη Συρία. Και θα ήθελα να παρακαλέσω εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της ε, ε, Επιτροπής είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για την Πολιτική Ασφάλειας ε, να πάρει το λόγο ο κύριος Βίλι Σεβδάλ. Παρακαλώ. Thank you very much, ε, Mr. President. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τις πιο πρόσφατες ε, δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Συρία εξ ονόματος της υπάτρες ε, προσώπου Άστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί την αύξηση της βίας στην Συρία. Έφτασε η ώρα να μιλήσουμε με μία φωνή και να σταματήσουμε ε, τις εξελίξεις αυτές στην Συρία για να υπάρχει μια δημοκρατική εξέλιξη. Χρειάζεται δράση των Ηνωμένων Εθνών. Απογοητευόμαστε πολύ, όπως και όλοι εσείς, από τις πρόσφατες αποτυχίες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να υιοθετήσει ένα ψήφισμα λόγω της αντίθεσης της Ρωσίας και της Κίνας. Το περασμένο Σάββατο η Πάτια Πρόσωπος είπε για άλλη μια φορά στη ότι συνεχίζει την υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, δημοκρατικών προσπαθειών και θα φροντίσει να αναλυφθούν οι σχετικέ ευθύνες. Η κρίση της Συρίας εξακολουθεί να παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων θα την ξανασυζητήσουν στις 27 Φεβρουαρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε στο πλευρό του Συριακού λαού και η ύπατη εκπρόσωπο, εξακολουθεί να αυξάνει την πίεση στι ε, αρχές ε, της ε, Συρίας σε πολλά επίπεδα. Η κύρια προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει αυτή η διάπλωση της βίας. Σύμφωνα και με τα σχέδια του Αραβικού Συνδέσμου είναι πάρα πολύ σημαντικό να απελευθερηθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και να επιτραπεί στα ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε ανεξάρτητους να πάνε στη Συρία. Για την επίτευξη αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στενά σε συνεργασία με τον Αραβικό Σύνδεσμο και με άλλες χώρες για να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Η ύπατη εκπρόσωπος τόνισε τον βασικό ρόλο της ηγεσία του Αραβικού Συνδέσμου σε διπλωματικό επίπεδο η Κάθριν Έστον συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα για το θέμα των βημάτων που πρέπει να αναλυφθούν και να συζητήσει τις πολιτικές προσπάθειες που αναλαμβάνει και ο, ο Αραβικός Σύνδρομος για να, λυθεί, για να λυθεί το πρόβλημα. Συζήτησε επίσης με τον Βανκιμούν, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με τον Τάβι Τσούπλο, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικό και άλλους ηγέτες που έχουν τους ίδιους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χαιρετίζει την προσπάθεια πολλών χωρών να αυξηθεί η διεθνής πίεση στην Συρία. Λόγω της ανόδου της βίας κατά του πληθυσμού της Συρίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αποσύρει την αποστολή της ε, εκεί. Εξτάττει το θέμα μιας ειρηνευτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτήρηση της εφαρμογής της ανακοπής του πυρός. Επίσης θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παλιότερα ψηφίσματα του Αραβικού Συνδέσμου και αναφέρεται ότι στι 26 Φεβρουαρίου θα πρέπει αμέσω να γίνει συζήτηση στην Ισία για το θέμα αυτό. Χαιρετίζουμε τι εξελέξεις αυτέ. Αυτή η συνάντηση τίνιδα θα επιτρέψει τη δυνατότητα δημιουργία ε, διεθνού συνένεση για τη Συρία και την προώθηση ε, προτάσεων για να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί η διέξοδο από την κρίση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΥΠΑΤΕ εκπρόσωπος θα παίξουν ένα ενεργό ρόλο. Η Πατεκπρόσωπος επίσης πρότεινε την ε, εμπειρονομοσύνη της Ένωσης όσον αφορά το θέμα των κυρώσεων και προτείνει να παραμείνει σε στενό διάλογο με τις ομάδες αντιπολίτευσης. Συνεχίζουμε να αναζητούμε την υποστήριξη των εταίρων μας, ότως ώστε να μπορεί να επανέλθει το Συμβούλιο Ασφαλείας στο θέμα αυτό και να συμφωνηθεί ένα καλό ισχυρό ψήφισμα για τη Συρία. Η πρόσωπος Παρουσιάζει το θέμα στα μέλη του Συμβουλίου Αυστραλία, ε, Ασφαλείας και τους άλλους εταίρους για το θέμα αυτό. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία και την Κίνα είναι σαφές. Δεν θα πρέπει να βρεθούν στην εσφαλμένη μεριά της ιστορίας. Η διεθνή κοινότητα έχει την ευθύνη να σταματήσει το καθεστώς να σκοτώνει τον πληθυσμό. Την περσμένη εβδομάδα στη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η μεγάλη πλειοψηφία καταδίκασε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς της Συρίας. Η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι θα πρέπει η Συρία να πληρεί τους προϋποθέσεις για την προστασία των, ε, του πληθυσμού και να μην συνεχίζει με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πράττει. Θα πρέπει επίσης στην επόμενη συνεδρίαση να ληφθούν σημαντικά βήματα για την Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει το άχθος του ε, συριανικού πληθυσμού και να προχωρήσει στην ε, χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας μερή συνεργασία με το καθεστώς της Συρίας έχει διακοπεί αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν εξακολουθεί να υποστηρίζει σχέδια προς όφελος μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων της ε, κοινωνίας των πολιτών και προτροπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και των Παλαιστινιών προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση μέσω των αποστολών των κρατών μελών όπως μας το ζητά και η, Συριακή, η Αντιπολίτευση. θα πρέπει να καταδεχθεί σε καθαρά ότι δεν επιτρέπεται το καθεστώς να καταστέλει το πληθυσμό κατά τέτοιον τρόπο αδημορητή. Στενή συνεργασία μεταξύ των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δαμασκό λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή και όσον αφορά για τα σχέδια δευτέρας ε, γραμμής. Τέλος, εξουσιασματικό όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει τη συνεργασία με τις ε, Συριακές Ομάδες Αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να ενδυναμωθεί ο συνονιστός της και να βρεθεί μία οδός προς τα εμπρός, ούτως ώστε να πιστεί ο πληθυσμός εκεί όσον αφορά την ε, δυνατότητα ειρηνικής μετάβασης. Η ύπατη εκπρόσωπος προσέφερε την, ε, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες αυτές ούτως ώστε οι ομάδες της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να συνεργαστούν προς μια ειρηνική μετάβαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ε, τέος δήλωσή σας στο παρελθόν το ψηφίσματα που γίνονται εδώ στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο βοήθησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, σχηματίσει την πολιτική της ε, για τη Συρία. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση της Συρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ρόλο να παίξει ούτω ώστε ο πληθυσμό τη Συρίας να μην εγκαταλειφθεί στη μοίρα του. Η ύπατη εκπρόσωπο έχει αναλάβει την υποχρέωση να συνεχίσει μαζί σα κοινέ προσπάθειε για να υποστηρίξει τον Αραβικό Σύνδεσμο και να υποστηρίξει τι προσπάθειες που γίνονται. Θα υπάρξει μια συνάντηση σχετική στην Ουάσιγκτον στα τέλη τη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόφταλ. Ε, περνάμε τώρα στου ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων και ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Σαλαφράγκα εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να πάρει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τρεις παράγοντες αλληλεξαρτώμενοι ε, βρίσκονται σε εξέλιξη με την κρίση στη Συρία. Πρώτα απ' όλα ψυχρός πόλεμος μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν αυτή τη στιγμή Κάτι που το βλέπουμε ε, σε πολλές περιπτώσεις και συγκεκριμένα τώρα το βλέπουμε στη Συρία. Επίσης, ε, κατάσταση ντόμινο σε ό,τι αφορά την αρινή την Αραβική Άνοιξη και επίσης ε, η δραστηριοποίηση Κίνας, Ρωσίας και άλλων παραγόντων για να καλυφθεί το κοινό που έχουν αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, ακούσαμε τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΠΑΤΗ πρόσωπος, αναστολή τη συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια, σχέδιο έκτακτης ανάγκη, ενίσχυση των κυρώσεων στο προσεχέ ε, συμβούλιο τη 27 η στήριξη των πρωτοβουλίων του Αραβικού Συνδέσμου. Τουλάχιστον μια πιο συντονισμένη απάντηση βλέπουμε, ε, διπλωματικά πιο αποτελεσματική από τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς καμία Καμία από τις αποφάσεις ε, δεν είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί βραχυπρόθεσμα η απαράδεκτη βία, ε, θύμα της οποίας είναι ο πληθυσμός της Συρίας. Όλοι είμαστε απογοητευμένοι. Σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την απογοήτευσή του. Πρόσφατα ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είχε πει πόσο απογοητευμένος είναι και με το βέτο της Κίνας Στη Γενική Συνέλευση τώρα συζητείται πρωτοβουλία του Κατάρ και της Σαουδική Αραβίας ε, για την επικύρωση της συμφωνίας αυτής που ξέρουμε όμως ότι δεν έχει κάποια δεσμευτική ισχύ. Τι μπορούμε να κάνουμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Θα μπορούσαμε σίγουρα να αυξήσουμε τις πιέσεις ε, προ την ε, Ρωσία και προ την Κίνα. Και είχαμε δύο δυνατότητε, δύο ευκαιρίε. Η πρώτη ήταν η επίσκεψη ε, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Κίνας, της ΕΕ, τον δέχτηκαν με όλες τις τιμές και η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ήταν η δεύτερη ευκαιρία που μόλις έγινε. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις μας με την ε, Συριακή Αντιπολίτευση, τους αντιφρονούντες από τη Συρία και να δούμε πώς ε, μπορούμε αυτόν τον ανθρωπιστικό διάδρομο που μας, έχει που μας έχουν ζητήσει οι αντιφρονούντες να τον εξασφαλίσουμε. Τις ερωτήσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, Υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου μας προβληματίζουν και εμάς. Δηλαδή, μέχρι πότε θα μείνουμε άπραγοι και απαθείς μπροστά στη βία που βλέπουμε να βιώνει ο λαός της Συρίας αυτή τη στιγμή. Ποια είναι τα όρια της, αντοχής, της ανοχής μας όταν βλέπουμε ε, μετά από οποιαδήποτε προθεσμία και πρωτοβουλία να παραμένει το καθεστώς ε, και να ματοκυλάει τη χώρα του και το λαό του. Ε, Θέτω αυτό το βασικό λοιπόν θεμελιώδες ερώτημα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαλαφράγκα, ήθελα τώρα να παρακαλέσω την κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι το το ψήφισμα που κάνει το Κοινοβούλιο για τη Συρία. Και θα έλεγα ότι η προστιθέμενη αξία αυτής της ε, ε, αυτού του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη και τις διπλωματικές προσπάθειες ή έστω μία από τις προσθέμενες αξίες είναι ότι λέμε στο Συριακό λαό έστω και αν τίποτα δεν γίνεται δεν σας ξεχνούμε, δεν λησμονούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι το ψήφισμα αυτό δεν απαντά ε, στα πιο σημαντικά ερωτήματα, ε, δηλαδή στο τι κάνουμε, τι πρόκειται να κάνουμε, ποιε είναι οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουμε, ποια είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Είναι αυτή η ερώτηση που με δάκρυα στα μάτια μου έκανε σήμερα το πρωί ένα μέλος του Συμβουλίου της ε, Συρίας, ε, του Εθνικού Συμβουλίου ε, που μου μίλαγε για τους νεκρούς, για τα βασανιστήρια και μου, δεν μου ζήτησε ούτε χρήματα, δεν μου είπε ούτε τι θα μας στείλετε, είπε θα μας βοηθήσετε, θα κάνετε κάτι και εγώ αναγκάστηκα να του πω ότι αυτό δεν αναφέρεται ούτε καν στο ψήφισμα γιατί δεν έχουμε τις σωστές διάβλους επικοινωνίας, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, δεν ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα. Μα ποια είναι αυτή η αξιοπιστία που περνάμε προς τον λαό της Συρίας. Αυτό περιμένουμε. Δεν στρέφομαι ούτε προς τον ένα σας ούτε προς τον άλλο. Ε, λέω απλώς τι θα κάνουμε και να πω για τον Μπασάρ Λάσαντ. Ε, μερικοί μεταξύ ημών πιστέψαμε πραγματικά και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το συριακό καθεστώς. Ε, θυμάμαι ότι ήμουν στο διαμέρισμα του Μπασάρε Λάσαντ που μου εξηγούσε ε, πώς θα πρέπει να αλλάξει η χώρα του και πώς έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της αλλαγής. Ε, μου έδωσε υποσχέσεις ε, για νέα συντάγματα. Πιστέψαμε τότε, εσφαλμένα προφανώς, τα, τις υποσχέσεις αυτές. Αλλά πραγματικά τα πράγματα τώρα πλέον έχουν ξεφύγει. Δεν συμφωνώ ούτε με τις εικόνες του ε, Σαντάμ Χουσέιν ούτε και με τις ε, εικόνες που είδαμε του Καντάφη αλλά παρόλα αυτά το φάσμα αυτό κρέμεται πάνω από το κεφάλι του. Θα πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος και εν πάση περιπτώσει εμείς εδώ θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Ζητώ προς, από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις θέσεις αυτές και να ξεκινήσει πλέον να γίνεται κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ντεκεζέρ. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, πρόεδρο κύριο Φερχόφσταντ. Ευχαριστώ πολύ. Χθε ε, η κάθε Άστον μου έστειλε μια επιστολή για να μου πει ότι ο εξ τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση τη ομάδα επαφή στην την Ισία στις 24 Φεβρουαρίου. Καλό αυτό, αλλά για να είμαστε ειλικρινεί αγαπητοί συνάδελφοι, τι στρατηγική εκεί πάμε να υπερασπιστούμε. Πρέπει να σα πω, κύριε Υπουργέ, δεν άκουσα κάτι πάνω στη στρατηγική Μα αναφέρατε τα αιτήματα του Αραβικού Συνδέσμου, αλλά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι στρατηγική έχει. Τι στρατηγική έχει απέναντι στη Συρία προ το παρόν. Είμαστε στη μέση αυτή τη ε, κρίση. Έχουμε ε, τα προβλήματα στη Χόμ. Δεύτερη Σρεμπρένιτσα, πραγματικά. Και μιλάμε για πόλεμο. Δεν μπορούμε, μα λέτε να μην αρθρώσουμε τη λέξη πόλεμο, μα για πόλεμο πρόκειται. Πρέπει να μα πείτε ποια στρατηγική έχουμε απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν αρκεί να μας λέτε ότι θα είμαστε στην Τινησία στις 24 του μήνα. Τι θα τους πούμε, ποια είναι η θέση μας για τα βασικά ζητήματα, τα οποία είναι επί τη ουσία Είμαστε υπέρ ανθρωπιστικής παρέμβασης στη Συρία για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών και ζωνών απαγόρευσης πτήσεων ε, στα σύνορα με την Τουρκία και την Ιορδανία, να έχουμε διαδρόμους. Εκεί είμαστε υπέρ, ναι ή όχι αυτή της πρότασης. Και νομίζω ότι είναι κάτι απολύτω απαραίτητο, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται γενοκτονία στη Συρία. Αυτό είναι. Και αν δεν το σταματήσει η διεθνή κοινότητα θα συνεχιστεί. Και τι θα κάνουμε στην ε, αντιπολίτευση και στον ε, ε, στρατό τους, θα τους δώσουμε βοήθεια ηλική. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστούν όπλα. Ε, στρατό, ίσως όχι στρατό γιατί αυτό μπορεί να το κάνουν ενδεχομένω ε, οι ε, συναδελφοί μας από τον αραβικό σύνδεσμο αλλά εγώ σας ρωτώ υλικό, εξοπλισμό που χρειάζονται αυτή την, τον τεχνικό εξοπλισμό μπορούμε να τους προσφέρουμε, τον χρειάζονται και δεύτερο ερώτημα, τι γίνεται με το καθεστώς των κυρώσεων από την αρχή γνωρίζουμε ότι ο κατάλογος μας ήταν πάρα πολύ μικρό. τουλάχιστον 200 οικογένειες ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο ε, καθεστώς του Άσαντ. Αρχίσαμε με 20, με 30, με 40, έτσι πάμε. Δεν μιλάω για οικογένειες και απλά για άτομα. 30-40 μιλάω. Τι θα γίνει, θα αγγίξουμε τις 200 μεγάλες οικογένειες. Και το επόμενο ερώτημα είναι αυτό που είπε και ο κύριος Σαλαφράγκα. Με τη Ρωσία, με την Κίνα, τι κάνουμε. Έχουμε ίσως τη δυνατότητα κάτι να πούμε και γι' αυτό σε αυτές τις δύο χώρες. Είχαμε την αποστολή, την αντιπροσωπεία στην Κίνα. Και τι τους υποσχόμαστε αυτή τη στιγμή, τους υποσχόμαστε το καθεστώς ε, της ε, χώρας ελεύθερης οικονομίας, όταν αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Δεν το νομίζω. Πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να πούν ναι σε παρέμβαση στη Συρία. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Θέλω από εσάς να ακούσω πραγματικά ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας είπατε πριν από λίγο. Θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών στις 27. Μας το είπατε αυτό. Τρεις μέρες μετά τις 24 δηλαδή. Πριν πρέπει να συνεδριάσετε. Πριν πάει η κυρία Άστον στην Τινησία. Μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη με αυτά που έχουμε κάνει, όπως στην περίπτωση της Λιβύης για παράδειγμα. Έχουμε μία μπλε κάρτα. Από τον κύριο Ντέβα δέχεστε την μπλε κάρτα αυτή. Κύριε Ντέβα, παρακαλώ. Δεν ακούγεται ο κύριος Ντέβα. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Ντέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσετε κύριε Βουλευτά ότι το 2006 στα Ηνωμένα Έθνη ξεκινήσαμε αυτή την ε, διαδικασία διαδικασία ε, ε, ανάγκη σε ε, προστασίας και ευθύνης προστασίας. Δεν βλέπω αυτή την θέση. Ποια είναι η ευθύνη προστασίας χρησιμοποιώντας το εργαλείο των Ηνωμένων Εθνών το οποίο δημιουργήσαμε. Θα συμφωνήσει ο φίλος μου εδώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και το Συμβούλιο αυτές τις ιδέες, αυτή την αντίληψη της ευθύνης προστασίας και ότι θα πρέπει να... Την έχουμε χρησιμοποιήσει στη Σιέρα και σε άλλες ε, χώρες. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε την τύχη των ε, αθώων ανθρώπων. Ναι, αυτή όμως είναι ερώτηση προς το Συμβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κλέψω όλο από το Συμβούλιο, αν θέλετε σας απαντώ. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, άποψή μου είναι ότι αν συμφωνούμε στην ομάδα επαφή, επαφής, ε, μπορούμε να αλλάξουμε τη διαδικασία. Δηλαδή, εάν ε, η Κίνα και ε, η Ρωσία δουν ότι όλοι οι υπόλοιποι και η ομάδα επαφή είναι απολύτω αποφασισμένοι να κάνουν κάτι έτσι ώστε να βοηθήσουν τον κόσμο, τότε νομίζω ότι θα αλλάξει η κατάσταση αυτή που είδαμε τον τελευταίο χρόνο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφεί. θα πρέπει να δείξουμε ότι πραγματικά ε, προστατεύουμε του ανθρώπου αυτού και ότι πηγαίνουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ελέν Φλότρο, εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως πιστεύω ότι εδώ πια δεν πρέπει να μιλάμε για ε, καταπίεση του λαού, αλλά για μια γενοκτονία πλέον του καθεστώτος ε, Μπασάρ να δει κανεί ότι τα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή είναι, ε, είναι σκηνέ απαγωγών, ε, τόποι βασανιστήριων, είναι κολαστήρια. Ξέρουμε ποιος είναι περίπου ο αριθμός των νεκρών, δεν είμαστε βεβαίω σίγουροι το είπε και το είπαν και τα Ηνωμένα Έθνη, πρόκειται για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έχει δίκιο η κυρία Ντεκεζέρ σε όσα είπε προηγουμένως. Θα πρέπει όλα αυτά τα εγκλήματα ε, να συζητηθούν ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης. Ε, βεβαίως θα πρέπει εδώ να μιλήσουμε ε, και για την κοινωνία των πολιτών της Συρίας, για, την, για τον θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο έχουν καταφέρει να οργανωθούν οι αντιφρονούντες παρόλες τις δυσκολίες και παρά τις, την απίστευτη κατάσταση που επικρατεί, καταφέρουν να επικοινωνούν, να, αντα, να, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ε, ε, έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν πρόχειρα νοσοκομεία, να περιθάλπτουν τους αρρώστους, τους, τους τραυματισμένους. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε ε, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ενταθεί η προστασία, η διακίνηση φαρμάκων, τροφίμων μέσα από αυτές τις ε, παράνομες διάβλους. Να βοηθήσουμε και εμείς. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς που με κίνδυνο της ζωής τους λαθρέα ε, διακινούν αυτά τα είδη, τρόφιμα, φάρμακα κλπ. Πιστεύω ότι βεβαίως θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι κυρώσεις και ότι οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε την σωστή τους εφαρμογή. Και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναρωτηθούν πώς ένα πλοίο γεμάτο όπλα έφυγε από ένα λιμάνι κυπριακό για να πάει στη Συρία έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα κατά του λαού της Συρίας. Θα πρέπει να στηρίξουμε και τον Αραβικό Σύνδεσμο. Πολύ προσεκτικά φυσικά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος είναι ένα συνοθήλευμα αντιφατικών και αντιλεγόμενων συμφερόντων αλλά παρόλα αυτά τούτη τη στιγμή ε, θα πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να βασιστεί λίγο και στον αραβικό σύνδεσμο όμως να πει και συγκεκριμένα τι θέλει. Βεβαίω οι φίλοι τη Συρίας που θα συναντηθούν στην Τινησία είναι κάτι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η δικιά μα θέση. Η θέση μα απέναντι σε ένα λαό ο οποίο αντιστέκεται, ο οποίο προσπαθεί να ε, κερδίσει την ελευθερία του. Ξέρουμε ότι ε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιόνια σε μια διεθνή κακέρα όπου κάθε μια κίνηση που κάνουμε, κάθε μια κίνηση που γίνεται τροποποιεί εντελώς τη θέση όλων των άλλων πιονιών στη κακέρα αυτή. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα διακυβεύματα εδώ. Αυτή η συνεδρίαση λοιπόν της 24ης θα πρέπει να απομονώσει τις χώρες οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να στηρίζουν ε, ε, τη Συρία. Δεν είναι μόνο η Κίνα, δεν είναι μόνο η Ρωσία, είναι και η Αλγερία. Θα πρέπει να απομονωθεί ο Ασάντ. Αυτό θα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο βοήθεια. Και θα πρέπει να στηρίξουμε το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να έχει τα μειονεκτήματά του, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα πολιτικό διάλογο πολιτικό διάλογο με την μελλοντική πολιτική κυβέρνηση της Συρίας. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τάνοκα, του συντηρητικούς βλέπουμε να γίνονται αποτροπιαστικά πράγματα στη Χόμς ε, και πρέπει να το καταδικάσει η, ε, η διεθνής κοινότητα ε, για το ψήφισμα το οποίο καταδίκαζε τις γενοκτονίες και τα, το οποίο δεν ψήφισαν Ρωσία και είναι και αυτό ντροπιαστικό θα πρέπει να αποσύρει ο Άσαντ τα στρατεύματά του από όλε τι πόλει τη Συρία, να παράσχει πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και να δρομολογήσει εκλογέ. Ε, ο ρόλος της Τουρκίας για την ε, υποδοχή προσφύγων είναι πάρα πολύ θετικός. Ο Αραβικός Σύνδεσμος προσπαθεί να τερματίσει τη βία και, αυτός πρέπει, και οι προσπάθειές του πρέπει να τύχουν ε, συγχαρητήρων. Πρέπει χωρίς καθυστέρηση η Συρία να αναγκαστεί να εγγυηθεί την προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών, να εγγυηθεί μεταξύ άλλων την ελευθερία έκφρασης. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι δυνατό όσο είναι ο Άσαντε στην εξουσία γιατί αυτός έχει οποιαδήποτε, την ευθύνη μάλλον για οποιαδήποτε κλιματική ενέργεια για ε, του ε, στρατού και ε, πολλών συγκεκριμένων μονάδων του, του στρατού θα πρέπει να παρετηθεί. Για το συμφέρον του λαού, ο κύριος ζήτησε να παράσχουμε στρατό, αυτό είναι επικίνδυνο. Ε, δεν ξέρουμε τι ρόλο διαδραματίζει και η τζιχάντ. Ε, δεν ξέρουμε πώς υπάρξει τελικά ένας πόλεμος με το Χεσμπολάχ και το Ιράν που δίνουν όπλα στο Μπάθ και ε, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία να δίνουν όπλα σε άλλες μειονότητες. οι χριστιανοί, οι Δρούζοι, οι Αλεβίτες, όλοι αυτοί να αναγκαστούν να, μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και αν δεν εξασφαλίσουμε ίσω και μια ζώνη απαγόρευση των πτήσεων ή μια ελεύθερη ζώνη στα σύνορα τη Τουρκία, δεν μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Είναι όλα ρευστά. Πρέπει όμω ε, επιγόντω να υπάρξουν και άλλε κυρώσει στο καθεστώ τη Δαμασκού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Ε, Ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βίλι Μέγερ από την Ευρωπαϊκή Αριστερά για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ομάδα μου θα είναι κατά, ριζικά κατά οποιασδήποτε στρατιωτική εξωτερική επέμβαση για την επίλυση τη κρίση. Είμαστε κατά και στην επιχείρηση στη Λιβύη και γνωρίζουμε ε, τι τέλο είχε ο δικτάτορα Καντάφη. Πλήρωσε τα εγκλήματά του από την ε, ε, με μέσω μιας εξωτερικής ε, στρατιωτικής παρέμβασης που και αυτό όμως ήταν έγκλημα. Θα είμαστε λοιπόν εντελώς αντίθετοι με οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση. Και μας φαίνεται περίεργο, μας έδωσε και μια πληροφορία υπουργό, η οποία είναι σωστή σε ό,τι αφορά την ανάγκη να πάψει η καταστολή του καθεστώτος ε, του Ασάντ, γιατί σίγουρα αυτό πρέπει να τερματιστεί. Αλλά ε, δεν μιλήσατε για τη Τζιχάντ. Υπάρχουν Λιβανέζοι, ε, υπάρχουν από τη Σαουδική Αραβία ε, άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν, ζητούν από τους λέοντες της Συρίας να αντιδράσουν. Ε, από τα σύνορα περνάνε όπλα και από τα σύνορα της Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει και το τσιχάντ να το σταματήσουμε. Κύριε Μάγερ, ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέλντερ από το EFT παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η εικόνα ενός εμφυλίου πολέμου έγινε πια πραγματικότητα στη Συρία. Έλεγαν ότι κανένας δεν μας προστατεύει, κανένας δεν βοηθάει. Υπάρχουν εθνοτικές ε, διαφορές, ε, θρησκευτικές διαφορές σε αυτή τη χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται. Υπάρχει εναλλακτική στο καθεστώς που υπάρχει σήμερα. Η αντιπολίτευση δεν είναι ενωμένη ούτε πολιτικά ούτε στρατιωτικά. Πού θα βρεθεί λοιπόν η εναλλακτική λύση η βιώσιμη. Ορισμένοι λένε ότι η Αλκαΐδα είναι αναμειγμένη, υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Ε, ρωτούμε λοιπόν, θα υπάρξει μια διεθνής παρέμβαση και θα σταματήσει αυτή η αιματοχυσία στην Συρία. Εάν δεν υπάρχει εναλλακτική θα επιδιωτωθεί η κατάσταση. Άγερα, από τους σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Φαντάζομαι και εγώ να μπορέσω να μιλήσω ένα λεπτό παραπάνω όπως και η που προμίλησε. Όσον αφορά τις απαιτήσει για το διάθεση, όσο πάει και γίνεται πιο ριζοσπαστική. Υπάρχουν οι διάφορες διαδηλώσεις που είδαμε. Ε, οι εικόνες που είχαμε στο πλευρό δεν υπάρχουν όμως γιατί οι ακραίοι εξτρεμιστές απειλούν την ιστορική επανάσταση και εγώ κατάλαβα καλή Αλκαίδα σε ε, πόλεμο κατά του ΕΣΑΤ. είναι η θρησκευτική, ε, θρησκευτικό καθήκον των εξτρεμιστών να ρίξουν την ε, <clears throat> κυβέρνηση ΕΣΑΤ, να ξαναφέρουν τη Σαρία. Θα ήταν όμως καταστροφή αυτό για τις ε, δημοκρατικές ε, φιλελεύθερες δυνάμεις της χώρας. Αυτή θα ήταν η χειρότερη λύση. Ένας πραγματικός διάλογος με τον Ασάτ που βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο ήδη θα ήταν η καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Οπενμάγερ. Περνούμε τώρα στους υπόλοιπους γεγραμμένους ομιλητές. Θέλω πρώτα να παρακαλέσω τον κύριο Γιάννη Κασουλίδη να πάρει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κτρία αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, να ε, πάρει αποφάσεις ε, κατά του καθεστώτος Άσαντ μέσα από την ψήφο της Κίνας και της Ρωσίας καταλήγει σε έναν πόλεμο με πολλούς τραυματίες και νεκρούς, κυρίως μεταξύ των αμάχων και των γυναικοπαίδων. Πρέπει να καταδικάσουμε την κατάσταση αυτή ε, γιατί υποτίθεται ότι ο κύριος Λαυρόφ ε, είπε ότι κινήθηκε με τον τρόπο αυτό έτσι ώστε να αποφευχθεί ο εμφύλιος πόλεμος αλλά δεν είναι δυνατόν ε, να αποφευχθεί τελικά ο εμφύλιος πόλεμος γιατί ξέρετε ότι οι απελπισμένοι άνθρωποι παίρνουν εν τέλει απελπισμένα μέτρα και επομένως οδηγούνται προς τον εμφύλιο πόλεμο αλλά ξέρουμε ότι και το καθεστώς ε, Άσαντ έχει ένα λόγο ε, που φέρεται με τον τρόπο αυτό γιατί προσπαθεί να κρατήσει την καθεστική ατάξη όσον αφορά τους Χεσμολά ε, και την Τζιχάτ στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να δούμε την κατάσταση μονάχα σαν μια εσωτερική διαμάχη. Θα πρέπει να στηρίξουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως τα οι ανθρωπιστικές ε, ανησυχίες ε, δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίζουν καταστάσεις και πολιτεύματα και το μόνο που θα πρέπει να μας ε, ενδιαφέρει είναι η προστασία των αμάχων πολιτών. Δεν μπορούμε να μείνουμε τα χέρια δεμένα σε, μια σε ένα τέτοιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και σε μια τέτοια αιματοχυσία. Βεβαίω θα πρέπει να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες του Αραβικού Συνδέσμου καθώς ε, και την ε, συνεργασία επιτόπου μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και Αραβικού Συνδέσμου. Ε, ζητούμε από την ύπατη εκπρόσωπο να πάρει περιοριστικά μέτρα, να προτείνει επομένως περιοριστικά μέτρα και να λάβει συγκεκριμένη θέση αποκλείοντας και τις χώρες οι οποίες δεν θέλουν να μπει ένα τέλος σε αυτήν την απίστευτη καταπίεση. Δεν είναι δυνατόν. Η κυβέρνηση πατρός Άσαντ, καθώς επίσης και οι κυβερνήσεις των αντιστοίχων χωρών δεν επιβίωσαν, δεν θα επιβιώσει ούτε αυτή η κυβέρνηση. Άννα Γκόμες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την αλληλεγγύη του προς το λαό της Συρίας που αποφασιστικά ανθίσταται όσο καλύτερα μπορεί στο καθεστώς του Μπασάρ Ελάσαντ που έχει βομβαρδίσει πόλεις, έχει βασανίσει παιδιά. Οι συναντήσεις σε επίπεδο ΟΗΕ καταδικάζουν το καθεστώς ε, του Άσαντ, του ζητούν να σταματήσει τις ε, φρικαλαιότητες κατά του λαού του. Είναι σαφές ότι οι ΣΥΡΙ θέλουν να ε, φύγει από την εξουσία, να παρετηθεί και ο Άσαντ αλλά και οι συνεργάτες του θα πρέπει ε, να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους ε, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον Αραβικό Σύνδεσμο και άλλους ε, προαγωνιστές της ευρύτερης περιοχής. Θέλουμε να υπάρξει εκεχηρία, πρέπει να ανοίξουμε διαδρόμους για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια, για να βοηθήσουμε τη χώρα να προχωρήσει προς τον εκδημοκρατισμό. Χρειάζονται υλικοτεχνική ε, υποστήριξη ε, και βλέπουμε ότι και χώρες όπως η Τουρκία ε, προτείνουν βοήθεια. Θα πρέπει να στηρίξουμε το λόγο της Συρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να θέσει ενώπιον των ευθυνών του στη Ρωσία και την Κίνα γιατί ήταν επωνίδιστη η στάση τους απέναντι στα άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας όταν τελικά και απέτρεψαν το Συμβούλιο Ασφαλείας από τον εκτελέσει το καθήκον του και δίνει ουσιαστικά έτσι, ε, δίνουν αυτές οι δύο χώρες ε, στον Άσαντ ε, άδεια για να σκοτώνει το λαό του. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ρωσία ξεκολουθεί να πουλάει όπλα στον Άσαντ. Οι Οαχάμπης επίσης παρέχουν όπλα στους ακραίους, στα ακραία στοιχεία. Προσπαθούν να προσταθεροποιήσουν την ευρύτερη περιοχή. Ο ΑΣΕΤ θα πέσει. Είναι ζήτημα χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως χρειάζεται ένα στρατηγικό όραμα ευθύ αμέσως για να δει και την μετά σαν εποχή πώς μπορεί να την προγραμματίσει από τώρα. Πρέπει να υπάρχει ενότητα βάση της εθνικής συμφιλίωσης στη Συρία να υπάρξει ένα δημοκρατικό σύνταγμα και να γίνουν σεβαστά όλα τα δικαιώματα και των αλεβιτών και χριστιανικών μειονοτήτων. Σάκη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρο. Είναι εύκολο να καταδικάζει κανένας ε, τους βιασμούς και τους ε, θανατώσεις σε αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί μια πραγματική λύση. Καμία λύση δεν είναι εύκολη. Το μέλλον δεν είναι βέβαιο, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια και να βλέπουμε τον πληθυσμό της Συρίας να ε, σφάζεται. Δεν έχουν νερό, ενέργεια, ε, φάρμακα. Είναι ανθρωπιστικό το πρόβλημα δηλαδή ένα, μια καταστροφή για την οποία είναι υπεύθυνο ο Ασά. Θα πρέπει να τον φροντίσουμε να σταματήσει. Ο πρόεδρο Περχόστατ αναφέρθηκε στι προτεραιότητες της ομάδας μας και θέλω να προσθέσω κάποια βήματα που μπορούν να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση άσχετα από τη στάση της Ρωσίας ή ε, της Κίνας. Δεν θα πρέπει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην επιβάλλουν το εμπάργο <clears throat> όπλων Πώς έφυγε ένα πλοίο με ρωσικά όπλα από την Κύπρο για να πάει στη Συρία. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείε δεν επιτρέπεται να εξάγουν ε, υλικό που χρησιμοποιείται για την εποπτεία επί των, ε, πολιτών. <clears throat> Γιατί επίσης όσον αφορά τα καύσιμα χρησιμοποιούνται για τα τάγκς που είναι στους δρόμους του Χόμς. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα προσέξουμε. Επίσης θα πρέπει να ε, γίνει σωστή ενημέρωση του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι απελάσσονται και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να μπορούν να ενημερώσουν. Κυρίε και κύριοι, δεν μπορούμε εμείς ε, να αξιολογήσουμε ακριβώς ε, τις καταστροφές εκεί, αλλά υπάρχουν αριθμικά στοιχεία για 7.000 νεκρούς και 7.000 νεκρού, κρατούμενους. Επίσης πείνα. Αυτοί είναι άνθρωποι σαν εμάς που υποφέρουν. Το ίμιση των πληθυσμών ε, εκεί είναι κάτω των 26 και θα πρέπει να ξέρουμε το μέλλον των ανθρώπων αυτών όταν προσασπίσουμε τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους. Πολύ. Η κυρία Ατού παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση είναι δραματική, αυτή η κατάσταση στην οποία υφίσταται ο Συριακός ε, λαός και δεν είναι δυνατόν να μείνουμε αδιάφοροι, ούτε να σιωπήσουμε μπροστά στα όσα κάνει ο Μπασάρ Ελάσαντ και το καθεστώς του. Θα πρέπει να εκφράσουμε έντονα την στήριξή μας ε, στον λαό της Συρίας που υποφέρει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταδικάσουμε, να καταγγείλουμε το βέτο ε, των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη. Θα πρέπει οι δημοσιογράφοι να έχουν τη δυνατότητα ε, να κυκλοφορούν ελεύθερα στο Συριακό έδαφος. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε τρόφιμα, αλλά κυρίως ιατρικό-φαρμακευτικό υλικό, το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή ούτε στη, κυρίως ε, στα νοσοκομεία ε, και στην Ήπεθρο δεν περνάει καμία ανθρωπιστική βοήθεια και δεν έχουν καθόλου φάρμακα. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ε, Συριακή αντιπολίτευση, ε, κυρίως ε, μέσω του Συμβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου της ε, Συρίας. Και θα πρέπει να στείλουμε τον Άσαντ, καθώς επίσης και όλους τους υπεύθυνους μακριά από τη χώρα και ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο ομιλητής είναι ο κύριος Καμίνσκι. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε σήμερα εκκλήσεις για διάλογο με τον πρόεδρο Άσαντ. Νομίζω ότι ο πρόεδρο Άσαντ έχει περάσει πλέον την κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλο διάλογο. Το αίμα αθώων, το αίμα παιδιών, τα οποία βασανίστηκαν στις φυλακές της Συρίας, ε, μας κάνει να μην μπορούμε πλέον να συνομιλούμε με τον πρόεδρο Άσαντ. Πρέπει να πούμε πολύ ξεκάθαρα εδώ στο σύμβολο της ελευθερίας και της δημοκρατίας ε, ε, σε αυτό το χώρο που είναι και σημαντικός για το λαό της Συρίας. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Άσαντ πρέπει να φύγει και πρέπει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη με μια τεράστια πρόκληση. Ένα τεράστιο ζήτημα τίθεται. Είμαστε ένας χώρος συζητήσεων, είμαστε ένα φόρουμ στο οποίο απλά γίνονται συζητήσεις ή μπορούμε να στηρίξουμε και να προσπίσουμε τις αξίες επί των οποίων ε, οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν. Ε, πρέπει να αντιδράσουμε και απέναντι στου εταίρου μα, στην Κίνα και τη Ρωσία. Πρέπει να του δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Ρωσία και η Κίνα θέλουν να συνεργαστούν μαζί μα και εμεί θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί του, τότε η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να σεβαστούν τι δικέ μα αξίε, τι αξίε που εμεί σεβόμαστε. είναι ο κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου για ένα λεπτό. Κύριε συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, διερωτήθηκαν δίκαια πάρα πολλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτέ τι ουσιαστικά μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτηση όμω είναι προ τον εαυτό μα. Αν συνάδελφοι είμαστε στη θέση των Επιτρόπων ή του Συμβουλίου, στην ίδια αδυναμία θα βρισκόμασταν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αυτό που πρέπει, διότι δεν κατάφερε να έχει κοινή βούληση, πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική και ουσιαστική δύναμη να εφαρμόσει αυτή την κοινή τη βούληση προ την κατεύθυνση του διεθνού δικαίου και διότι στη σύγκρουση τη συγκεκριμένη μεγάλων δυνάμεων πάνω από τη συρία η ευρωπαϊκή ένωση φαίνεται απλώ να παίρνει τη θέση υποστήριξη μέρου των μεγάλων δυνάμεων παρά να έχει δική τη θέση και δική τη δυνατότητα θέση και δυνατότητα εναρμόνιση με το δίκαιο των πολιτών τη συρία στη συγκεκριμένη περίπτωση άλλωστε αν δούμε ειλικρινά τι έγινε με την αραβική άνοιξη στι υπόλοιπε χώρε τη περιοχή, δεν νομίζω να οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι καταφέραμε να κάνουμε το σωστό. καταλήγω πω αν η ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει δική τη αξιοπιστία και ικανότητα υπεράσπιση του δικαίου τότε θα συνεχίσει να παραπέει μονίμω μεταξύ τη θέση παρέμβαση και τη θέση του απαθού παρατηρητή και τα δύο βλάπτουν τη συρία το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηγεωργίου. Ε, ο κύριος Προβέρα Φιωρέλο δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Ε, ε, Herr Kollege Μπροκ, Elmar Brock, Sie haben das Wort. Für Έχετε λόγο κύριε Μπροκ για τρία λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Η περιγραφή είναι σαφής νομίζω, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. η μόνη νομιμοποίηση για όσα εκεί είναι κάποια οικογένεια, ε, ε, κάποια, ε, ομάδα ανθρώπων θέλει να κρατήσουν την ισχύ στα χέρια τους. Οι οπαδοί του καθεστώσεως θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο Ασάντ δεν έχει μέλλον και θα πρέπει να φροντίσουν να αλλάξει το καθεστώς. Αυτό είναι η πιο σημαντική μέθοδος. Θα πρέπει να είναι σαφής η κοινή θέση της ε, κοινωνίας των εθνών. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει η Ρωσία που έχει μέχρι στιγμή αρνηθεί να βλέπει ε, τι πρέπει να κάνει για να προωθήσει την, ε, την ανθρώπινη πτυχή και να μην προσπαθεί μόνο να πουλήσει όπλα. Το σημαντικότερο είναι να συνεργαστούμε με τον Αραβικό Σύνδεσμο που την περασμένη Πέμπτη υπέβαλε το ψήφισμα στα Ηνωμένα Εθνή θα πρέπει να τύχει ευρεία υποστήριξη για να μπορέσει να προχωρήσει. Μου φαίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι η συνεργασία με την Τουρκία και με την Αραβικό Σύνδεσμο είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αυτό δεν θα πρέπει να είναι θέμα μόνο των δυτικών, είναι μια συνεργασία με ηγεσία του Ραβικού Συνδέσμου και με στενή συνεργασία με την Τουρκία. Αν μου επιτρέψετε να το ξαναδιατυπώσω, κύριε Σιγηρή, έχουμε εμπειρία από την Αίγυπτο, από τη Λιβύη και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει απαραίτητο διάλογο και με την αντιπολίτευση. Η κυρία Γκόμες το ανέφερε, αναφερθήκε στι γλώσσε τη μειονότητα. Θα πρέπει τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η ανεξαρτησία να μην καταπατούνται. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ, μετά δίωξη των ε, χριστιανών γιατί η κατεύθυνση που θα πέρει η χώρα αυτή θα είναι ισλαμιστική. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πλήρης υποστήριξη και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να μην υπάρχουν μετά ε, αδικίες από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να απομονωθεί ο ΑΣΑΤ στη χώρα του και να σκεφτούμε και τι θα γίνει μετά. Γιατί υπάρχουν και ορισμένε μειοψηφίε στο πλευρό του ΑΣΑΤ γιατί ελπίζουν ότι αυτό θα δώσει μεγαλύτερη σταθερότητα. Και θα πρέπει να φροντίσουμε οι εθνοτικέ και θρησκευτικέ ε, μειονότητε να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν ειρηνικά σε αυτή τη χώρα. Και θα πρέπει και τα θέματα να τα και από αυτή τη σκοπιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπροκ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Σαΐντ Ελ Καντράουι. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλοι είμαστε εγχωμένοι μετά από το βέτο της Κίνας και της Ρωσίας γιατί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η βία είναι ακόμα περισσότερη και κινδυνεύει ε, η βία να συνεχίσει για πάρα πολύ καιρό φαίνεται ότι οι όποιες κυρώσεις δεν προβληματίζουν καθόλου το καθεστώς Άσαντ. Όμως οι προσπάθειες πρέπει να συνεχίζονται και συνεχίζονται και από την πλευρά του Αραβικού Συνδέσμου και από την Τουρκία. Ε, είναι γεγονός ότι και κάποιες οικονομικές ε, κυρώσεις ε, θα υπονομεύσουν κάπως το καθεστώς. Αλλά βεβαίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να απομονώσουμε την κυβέρνηση του Μπασάρε Λάσαντ. Χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία που δεν επιτρέπουν στην διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την Συρία. Ε, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μας προβληματίζει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα κατάλογο με τις ε, διεθνείς, ας πούμε, εταιρείε ε, οι οποίες στηρίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη Συρία. Μπορούμε να στηρίξουμε επίσης τις μειονότητες, αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε σαφή και αξιόπιστο πολιτικό λόγο, αλλά και ένα σχέδιο έτσι ώστε να γίνει κατανοητό σε όλες ε, τις ε, μειονότητες ε, ότι θα εξαρτηθεί από τη στάση τους και η στάση που θα έχει η διεθνής κοινότητα απέναντί τους μετά την απομάκρυνση του Μπασάρε Λάσαντ. Θα πρέπει φυσικά να δουλέψουμε και με την Αραβικό Σύνδεσμο και με την Τουρκία έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως και το Ιράκ έτσι και η Συρία είναι ένα μοσαϊκό, όπως εκτός έχει ισχυρό στρατό και όπως η Λιβύη ο Άσαντ ε, σφαγιάζει τον ίδιο του το λαό. Ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτό τον πιο ισχυρό πονοκέφαλο, αν θέλετε, στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης είναι να μην κάνει λάθη πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι η αφετηρία. Πρέπει να είμαστε επίσης αξιόπιστοι και υπεύθυνοι. Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία μας, πώς μπορούμε να κάνουμε κηρύγματα στην Κίνα και στη Ρωσία όταν η Μέρκελ, η Άγγελα Μέρκελ μίλησε όπως μίλησε στην Κίνα Βλέπετε ότι και οι κυβερνήσει μας επιδοτούν ακόμη το σειρακό καθεστώ. Θα διαβάσετε στις ειδήσει, μπορείτε να τα δείτε στο ίντερνετ. Ούτε καταφέραμε να καταλήξουμε σε συνένεση για το άνοιγμα ε, ανθρωπιστικών διαδρόμων, να βοηθήσουμε τους ε, Σύρους ε, πρόσφυγες. Χρειάζεται αλληλεγγύη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει εάν θέλει ε, αυτό το παζλ της Ένωσης να το λύσει. Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα το οποίο έχουμε μπροστά μας έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία, όμως υπάρχει και ένα σημείο το οποίο δεν δέχτηκαν κάποιες πολιτικές ομάδες. Ε, υπάρχουν πολιτικές ομάδες οι οποίες αρνήθηκαν να περιληφθεί μια παράγραφος όπου αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε, ότι αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική επέμβαση. Ε, δεν ξεχνούμε τι συνέβη στη Λιβύη και δεν έχουμε βεβαίως και διασφαλίσεις ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα παίξει παρόμοιο ρόλο με αυτό που έπαιξε στην Λιβύη. Είναι γεγονός ότι η Συρία διαφέρει από τη Λιβύη, Λιβύη αλλά παρόλα αυτά ε, ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, ένας εμφύλιος πόλεμος στην Συρία θα μπορούσε ε, να διαχυθεί τελικά σε ολόκληρη την ε, περιοχή και επομένως το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε την θεμητή βούληση ενός λαού για ανεξαρτησία και για ελευθερία έτσι ώστε να ξανασχηματίσουμε τον πολιτικό χάρτη της περιοχής. Εμείς είμαστε δίπλα στο Συριακό λαό. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιάτσεκ Βλόσοβιτς. Για ένα λεπτό. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μου δώσετε το λεπτό του κύριου Προφέρα και να έχω δύο συνολικά λεπτά. Είναι δυνατόν, μπορώ να μιλήσω για δύο λεπτά, αφού ο κύριος Προφέρα δεν ήταν εδώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη ανάλυση για να δούμε τι γίνεται στη Συρία. 8.000 άνθρωποι περίπου έχουν χάσει τη ζωή της στη Συρία, εκ των οποίων αρκετές χιλιάδες ήταν παιδιά. Έχουμε 200.000 αγνοουμένους, 7.000 ε, κρατούνται στις φυλακές. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα δεν ε, παίρνουν βοήθεια οι Σύριοι, γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια ε, και τα φάρμακα δεν μπορούν να περάσουν γιατί τους πυροβολούν αυτούς που τα μεταφέρουν. Ε, υπάρχει υπάρχουν επιθέσεις από το πυροβολικό, δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς αυτούς που έχουν πυροβολήσει ελεύθεροι σκοπευτές. Βλέπουμε επίσης μισθοφόρους από το Ιράν να πολεμούν στη Συρία. Υπάρχει η Ρωσία η οποία εξακολουθεί να πουλά εξοπλισμό στη Συρία και επίσης υπάρχει αδιέξοδο στα Ηνωμένα Έθνη όταν ε, και υπήρξε βέτο κατά ενός ψηφίσματος. Ποια είναι η απάντηση κυρία Άστον, δια τους εκπροσώπου της, ε, είπε κάποια πράγματα και κάποιοι συνάδελφοί μας ε, μίλησαν. Ε, πρέπει να κλιμακωθούν οι κυρώσεις κατά του Συριακού καθεστώτος. Πρέπει να συνετιστεί η Ρωσία και η Κίνα και θα πρέπει να λογοδοτήσει στη Χάγη ο Άσαντ. Αλλά πρέπει, γιατί αυτά είναι για πιο μετά, πρέπει να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πώς θα σταματήσουμε τους θανάτους αθώων πρέπει να ε, αναγκάσουμε τον Άσαντ να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Πρέπει να πάψουν ε, οι πολιορκίες ε, των πόλεων, να ανοίξουν οι πολιορκημένες πόλεις. Βλέπουμε αύξηση των θανάτων. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να παράσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Μάριο Ντάβιτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτό το ημικύκλιο της δημοκρατίας ε, θα ε, καταδικάσει ε, τη στάση του Άσαντ και του καθεστώτος του που δολοφονούν αθώους πολίτες, κάτι που βλέπουμε καθημερινά. Θα πρέπει η Ευρώπη να μιλήσει με μια φωνή να μιλήσει ομόφωνα υπέρ του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, να καταδικάσει ε, τις αδιάκριτες ε, σφαγές ε, και την αιματοχυσία. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στο καθεστώς Άσαντ εφαρμόζοντας νέα περιοριστικά μέτρα. Θα πρέπει να πάψουν οι δολοφονίες, αλλά αυτό άλλωστε δεν μπορούμε καν να, να θεωρήσουμε ότι είναι υποδιαπραγμάτευση. Βέβαια θα χρειαστεί μια περίοδος μετάβασης στη Συρία. Όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν και όλες οι χώρες θα πρέπει να ακολουθήσουν ε, την ίδια ε, πορεία που δεν γίνεται. Είδαμε να απορρίπτονται δύο ψηφίσματα ε, στο πλαίσιο του, Συμβουλίου, του Ασφαλείας και έτσι συνεχίζεται η κατάσταση, συνεχίζονται οι σκοτομοί. Πρέπει να απομονωθεί η Ρωσία και η Κίνα που στηρίζουν το καθεστώς. Αλλά βλέπουμε ότι το καθεστώς, το πελπισμένο αυτό καθεστώ συνεχίζει να κρατιέται με το ζόρι στην εξουσία. Πρέπει η γενοκτονία αυτή να τερματιστεί. Έχουμε μείνει πίσω. Δεν έχουμε ακόμη σκληρίνει τη στάση μας. Πρέπει να στηρίξουμε τον Αραβικό Σύνδεσμο πιο συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις του και στην πρόθεσή του να στείλει και μία ε, δύναμη ειρήνευση στη χώρα. Θα πρέπει να στηρίξουμε ανεπιφύλακτα ε, και τις προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο ε, των Σύρων. Θα πρέπει διεθνής κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα για να τιμωρήσει τους ε, ε, εγκληματίες, ε, αυτούς που διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πρέπει να απαγορεύσουμε εμπορικέ συναλλαγέ Ευρωπαϊκή Ένωση με όλε τι ρωσικέ και κινέζικε επιχειρήσει που έχουν εμπορικέ σχέσει με τη Συρία. Θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθε. Επόμενη ομιλήτρια για 1,5 λεπτό είναι η κυρία Μαρίτα Ούλσκοκ. Herr talman! Eh, våldet regerar nu i Syrien. Κύριε Πρόεδρε, ε, υπάρχουν τεράστια προβλήματα με την ελληνική κυβέρνηση της ε, Συρίας. Ε, υπάρχουν πολύ ανησυχητικές μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων που ήρθαν και στο Στρασβούργο και μας μίλησαν που μίλησαν και μέρη εδώ έξω από το κτίριο αυτό, που ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Ξέρουμε και εμείς ένα μεταξύ τι γίνεται εκεί. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εκεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν αρκεί να δίνουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια όσο και αν είναι σημαντική αυτή. Ξέρουμε επίσης ότι ε, οι στρατιωτικές ε, πράξεις δεν είναι εναλλακτικοί. Το ψήφισμα του ΟΗΕ είναι βέβαια σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει μια, ε, ένα ευρύ πολιτικό μέτωπο στο οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα σταθούν ε, ο ένας δίπλα στον άλλον ούτως ώστε να δείξουν ότι είναι ισχυρή η διεθνής κοινότητα και αυτό για όλους, όχι μόνο για εκείνους που βρίσκονται στην Συρία. Είναι σημαντική η αλληλεγγύη. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση πάνω στη Ρωσία και στην Κίνα. Να ερευνήσουμε κάθε δυνατότητα για να αποτρέψουμε το στρατιωτικό, την, τον, το εμπόριο όπλων, αλλά δεν είναι λύση στρατιωτική λύση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Πολλές αλήθειες ακούστηκαν σήμερα εδώ και όλοι γνωρίζουμε ότι μέσω της συζητήσεως αυτής ε, μόνο λόγια μπορούμε να λέμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση εξ ολοκλήρου. Πάντως πιστεύω ότι είναι καλό που τουλάχιστον καταφέραμε να πούμε τις αλήθειες αυτές. Βεβαίως ε, συμφωνώ ότι δεν έχει καμία έννοια να κάνουμε διάλογο με, το καθεστώς ε, Μπασάρ Ελάσαντ, ε, θα, ούτε με τους εκπροσώπους της κυβέρνησής του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν τις προσταγές τους από τον ε, Πρόεδρο ε, και τελικά κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι αυτοί να βρεθούν ενώπιον του Διεθνούς ε, Δικαστηρίου. Βεβαίως θα πρέπει να καλέσουμε την Κίνα και τη Ρωσία έτσι ώστε να μην κλείσουν την οδό αυτή. Είναι μία οδός μια οδός εσχήνης ε, ε, που δεν είναι δυνατόν να ε, την αφήσουμε να συνεχίζεται. Είναι μια στάση η οποία πραγματικά θα πρέπει ε, να σταματήσει. Θα πρέπει να κάνουμε μια έκκληση ε, λοιπόν προς τις χώρες αυτές ε, και επίσης να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει αυτήν την αδύναμη έστω αντιπολίτευση που όμως υπάρχει να μπορέσει να καταλάβει η αντιπολίτευση αυτή ότι την στηρίζουμε. Όλες αυτές οι ομάδες ομάδες να καταλάβουν ότι με κάποιο τρόπο ε, τις ε, βοηθούμε. Να δημιουργήσουμε ενδεχομένως μια ομάδα φίλων της Συρίας στο Κοινοβούλιο. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μαρία Μουνίθ Λεορκίθα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβούλιο, κύριε Επίτροπε, χθε υπήρξε σύνοδο κορυφή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Τη ε, 15η Δεκεμβρίου είχε γίνει σύνοδος κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Τότε ε, είχε ξεκινήσει ε, την ματηρή καταστολή του δίτου του λαού το καθεστώς ε, του Άσαντ. Όμως, με τις δύο αυτές χώρες ξέρουμε τι έγινε, ξέρουμε ότι καταδίκασαν, μάλλον άσκησαν βέτο σε ένα ψήφισμα το οποίο θα καταδίκαζε τη στάση του καθεστώτος Άσαντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ότι έχει και αυτή κάποιο ρόλο να δραματίσει στη διεθνή σκηνή. Πρέπει να μπορεί να επηρεάζει τους συνομιλητές της, αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι στην ασημαντότητα. Η Ρωσία και εκείνο θα πρέπει να δεσμευτούν, να βάλουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω από την εθνική κυριαρχία. Δεν μπορεί ε, να υπάρχει ατιμορρησία. Ε, εμείς αποκλείουμε την στρατιωτική παρέμβαση, αλλά απαιτούμε τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Θα πρέπει να πάψει επίσης η καταστολή Σα Σας παρακαλώ λίγο ε, να είστε πιο γενναιόδωρος με το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να σταματήσουμε την καταστολή. Πρέπει να πάψουν οι πωλήσει όπλων, ε, να υπάρξει μαύρη λίστα και να μην στηρίζεται πλέον η κυβέρνηση. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Άνρο Ντάνζαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην ε, Συρία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο οδυνηρή πρόκληση που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα. Ε, το να βομβαρδίζει ο κυβερνήτης τον ίδιο το λαό με βαριά όπλα, ε, να τον κλείνει στις φυλακές και να τον βασανίζει, αυτό είναι πραγματικά εγκληματικές πράξεις. Είμαστε αγανακτισμένοι και αντιδρούμε, αλλά αυτό είναι πιο εύκολο από το να λαμβάνουμε συγκεκριμένη δράση. Ε, Βεβαίω το ενδεχόμενο στερεωτική παρέμβασης όπως στη Λιβύη είναι, ε, δεν ε, είναι ένα ενδεχόμενο και τα μέσα επέμβαση που έχουμε είναι πραγματικά πρέπει να το ομολογήσουμε πολύ περιορισμένα. Ο ίδιος ο πρόεδρος Μπροκ προηγουμένως αναφέρθηκε στον πιο ρεαλιστικό τρόπο αντιμετώπισης που είναι η, ο παραγωνισμό, που είναι η απομόνωση της Συρίας αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ενδιαφέρον ε, σχέδιο δράση. Ε, ε, όσον αφορά τη διπλωματική οδό, που είναι μια σημαντική διάσταση, Βεβαίω θα πρέπει εξ αρχή να καταδικάσουμε το βέτο των δύο χωρών και κυρίως να δώσουμε στις δύο χώρε αυτές να καταλάβουν ότι όχι μονάχα είναι απαράδεκτο, αλλά είναι και αδιανόητο, μη κατανοητό για τι υπόλοιπε χώρε μέλη. Ε, θα πρέπει ε, να στηρίξουμε και τον Αραβικό Σύνδεσμο, έστω και αν οι προτάσεις της δεν είναι πραγματοποιήσιμες βραχυπρόθεσμα. πέρα από την, από την πολιτική πρόκληση να στηρίξουμε ε, την, ε, να, στηρίξουμε την αντιπολίτευση ε, και να περιθωριοποιήσουμε χώρες όπως το Ιράν ή τη Ρωσία που στηρίζουν το καθεστώς Άσαντα θα πρέπει να προωθήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι δεοντολογική ηθική απέτηση αυτό. Θα πρέπει να προωθηθούν οι πρωτοβουλίες του Αραβικού Συνδέσμου και να σταματήσει αυτό το σκάνδαλο και της κατάστασης της Συρίας. Ε, επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Wolfgang Kreis, Kreis για ένα λεπτό. Εξότιμη συνάδελφοι, εδώ και ε, ναι, δέκα μήνες ο κύριος δι, καταδείχνει τη διεθνή κοινότητα σαν να είναι η αδύναμη, η λύθη υπάρχει μια πρόκληση για μαζικούς, ε, μαζικές θανατώσεις. Προσπαθεί να δημιουργήσει δεδομένα το καθεστώς αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά ένα πρέπει να είναι σαφές. Θα πρέπει οι κυρώσεις να ε, είναι πιο ισχυρές και δεν θα πρέπει να αρθούν ποτέ. Θα πρέπει να αρθούν μόνο όταν αυτό το καθεστώς υποχωρήσει και θα πρέπει οι υπεύθυνοι να ε, προσεχθούν στο Διεθνές Δικαστήριο στην Χάγη. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Θα πρέπει να ασκηθεί επίσης μεγαλύτερη πίεση στην Κίνα και στη Ρωσία. Και άμα εδώ όταν συζητάμε για το Μαρόκο και εμπορικές συμφωνίες έχουμε, έχουμε συζητήσεις επί συζητήσεων. Έχουμε εμπόριο όμως και με την Κίνα αλλά δεν συζητάμε τίποτα. Και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτούς τους ε, φόνους να συνεχίζονται. Ο ομιλητή, είναι ο κύριο Μίχαελ Γκάλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τι θα πρέπει να κάνουμε από κοινού τώρα. Όλοι ε, οι οποίοι έχουν ε, ευθύνη εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη θα πρέπει κάθε ευκαιρία να πιέζουν την Κίνα και τη Ρωσία να άρουν το φέτο τους αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει να κάνουμε και κάτι περισσότερο γιατί στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην ΩΣΑ θα πρέπει να δούμε ότι οι αρχές που ισχύουν εκεί ισχύουν και όταν δρούμε εκτός Ευρώπης. Ε, δεν επιτρέπεται η Ρωσία να εξακολουθεί να προμηθεύει όπλα σε, αυτή, σε αυτό το καθεστώς. Κύριε Πούτιν, κύριε Μεντιέβε, σταματήστε με την πρακτική αυτή ή αλλιώς θα θεωρείτε σαν και εκείνους τους εχθρούς που υπάρχουν γενικά στην ρωσική ιστορία. Γιατί δεν μπορέσαμε να αποσύρουμε τις εθνικές αντιπροσωπείες ε, από τη Δαμασκό. Ας ε, συνεργαστούμε στενά με την Τουρκία. Ας ε, μπορέσουμε να δράσουμε από κοινού, δημόσια. Παραδείγματος χάνει τη δημιουργία στρατοπέδων για τους πρόσφυγες στην τουρκική πλευρά των συνόρων. Ας φροντίσουμε να υπάρχει ένας διάλογος σε ψηλό επίπεδο και να κάνουμε κοινέ δηλώσεις προθέσεων για την εποχή μετά τον Ασάντ. Αυτές οι δηλώσεις θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και να λένε ότι όλοι οι Συροί, ακόμα και εκείνοι που ανήκουν σε θρησκευτικέ ή εθνοτικέ μειονότητες, έχουν ένα μέλλον. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει μια τέτοια Συρία στην οδό προ το μέλλον. Θα πρέπει επίση να φροντίσουμε σε περίπτωση που θα ε, πέσει αυτό το καθεστώς, θα υπάρχουν αλλαγές και στις γειτονικές χώρες. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και στη Λιβύη κάποια, στο Λίβανο συγγνώμη, θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Και θα πρέπει ήδη τώρα να κάνουμε έκκληση σε όλα τα μέρη εκεί να μην θεωρηθούν ότι μπορούν να ενθαρρυνθούν να εκμεταλλευτούν ένα κενό που ενδεχομένως θα υπάρξει στην Συρία. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, πρέπει να συνεργαστούμε για να διώξουμε τον Άσαντ και να ε, εκδημοκρατήσουμε τη Συρία. Και γι' αυτό απαιτούνται διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να στηρίξουμε τι ε, χώρε του Αραβικού Συνδέσμου στο σχέδιό του. Ε, πρέπει να συνεργαστούμε στενά με την Τουρκία, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρωταγωνιστή στην ευρύτερη περιοχή. Επίση, πρέπει να συνεργαστούμε με τη Ρωσία, όχι στο πλαίσιο του ΟΗΕ μόνο, αλλά και διμερό. Δηλαδή, μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία να υπάρχει συνεργασία. Τέταρτον, να συνεργαστούμε με τι δυνάμει τη αντιπολίτευση. πρέπει να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο εκδημοκρατισμού της Συρίας ε, για τη μετά τον Άσαντ εποχή. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε και με άτομα από το κυβερνόν κόμμα της Συρίας για να έχουμε ε, μια καλή μετάβαση. Το είδαμε και στο Ιράκ μετά το Σαντάμ. και βέβαια να αποτρέψουμε να μπουν Ισλαμιστές ε, στην εξουσία. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Συρία, η οδύνη, τα βάσανα του λαού δεν είναι κάτι καινούριο. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένο το ίδιο και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζουμε αυτά τα οποία ε, συμβαίνουν σήμερα στην ε, Συρία. Όλοι συμφωνούμε. Το να, στείλουμε ε, το να στέλνει μάλλον κάποιος και στρατό κατά του ίδιου του λαού είναι απόλυτα καταδικαστέο. Αυτό κάνει το καθεστώ που είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία στην Συρία. Όμω το ρωσικό και κινέζικο βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλεία επιδίνωσαν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στι δύο αυτέ χώρε για να αλλάξουν στάση. Θα πρέπει επίση να πάψουμε την εξαγωγή όπλων προ τη Συρία. Τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται κατά των διαδηλωτών. Ο Αραβικό Σύνδεσμο θα πρέπει να στείλει μια ειρηνευτική δύναμη, αλλά με την εντολή των Ηνωμένων Εθνών προσπάθειες του Αραβικού Συνδέσμου να στηρίξει την ε, αντιπολίτευση στη Συρία είναι ένα πρώτο βήμα. Ακούσαμε επίσης πόσοι έχουν σφαγιαστεί σε αυτή τη χώρα, πόσοι άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, πιστέψουμε ότι είναι δυνατή η δημοκρατική αλλαγή στη χώρα. Και υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο κυβερνοκόμμα που βλέπουν τα εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος του Συριακού λαού. Και ίσως αυτά τα άτομα θα ήθελαν να κάνουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Τα άρματα μάχη πρέπει να φύγουν από τους δρόμους. Οι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει να απελευθερωθούν. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει στον κόσμο. Για την ανθρωπιστική βοήθεια όμως, για να φτάσει στον προορισμό της, χρειάζεται και ανθρωπιστικός διάδρομος μέσω της Τουρκίας. Κάτι το οποίο προωθεί ως ιδέα ο Αραβικός Σύνδεσμος. Ο ανθρωπιστικό διάδρομος πρέπει να δημιουργηθεί για να σώσει τον κόσμο, τον κόσμο που ζει σε τραγική κατάσταση. Πρέπει να βοηθήσουμε τους τραυματίες και όλη την κοινωνία των πολιτών της Συρίας. Εγώ τώρα στην κυρία Κορίνα Κρέτσου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση στην Συρία χειροτερεύει από μέρα σε μέρα. Σφαγές γίνονται στις χώρες ε, όπου ο κόσμος ε, προσπαθεί μέσα από μια πλέον ε, ριζική μάχη να αντιμετωπίσει το καθεστώς μπασαρε Ελάσαντ. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει η κατάσταση αυτή. Θα πρέπει και τα Ηνωμένα Έθνη παρά το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των δύο χωρών θα πρέπει λέω να καταδικάσει σαφώς αυτή τη σφαγή των αμάχων. Θα πρέπει πρέπει και να στηρίξουμε τον Αραβικό Σύνδεσμο έτσι ώστε να είναι σαφής η πίεση προς ε, την κυβέρνηση της ε, Συρίας ε, θα πρέπει να βρεθούν έστω μέσω επιπλέον κυρώσεων λύσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το βήμα τον κύριο Πέτερ Στάζνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε τις απίστευτες ομότητες που λαμβάνουν χώρα στη Συρία τους τελευταίους 11 μήνες. Πάνω ε, από 500.000 ε, ε, Σύριοι έχουν χάσει τη ζωή τους. ο Αραβικός Σύνδεσμος ε, καταδικάζει ε, το καθεστώς ε, του Μπασάρ Ελάσαντ και τον καλεί να οργανώσει ελεύθερες εκλογές όπως έχει υποσχεθεί και στο παρελθόν. Στα Ηνωμένα Έθνη επίσης προσπάθησαν να περάσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας τέτοιου είδους κείμενα τα οποία όμως δεν πέρασαν λόγω του βέτο της Κίνας και της Ρωσίας υπογραμμίζω την ανάγκη περαιτέρω διπλωματική δράση, έτσι ώστε ε, να καταλάβει και η ρωσική κοινή γνώμη περί τίνο πρόκειται και να αλλάξει στάση τελικά η χώρα. Η ε, κυρία Άστον μίλησε με πολύ ισχυρό, ισχυρά λόγια ενώπιον του Κοινοβουλίου για, τον, ε, για την ανάγκη να συνταχθεί η Ρωσία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία στην χώρα αυτή Στηρίζω τις κινήσεις λοιπόν της Βαρόνης Άστον ε, καθώς επίσης ε, και όλων όσων αντιτίθενται σε αυτήν την ε, κυβέρνηση του πολέμου και της γενοκτονίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική πίεση στην ε, κυβέρνηση της Συρίας και θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να πιέζουμε την Ρωσία και την ε, Κίνα έτσι ώστε να μετακινηθούν από τις θέσεις τους. Τώρα το λόγο έχει ο, κυ... ο συνάδελφος κύριος Πάβελ Ζαλέσκι για δύο λεπτά. Ε, για άλλη μια φορά, έχουμε μια σημαντική συζήτηση για εξωτερική πολιτική στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και για άλλη μια φορά η κυρία Άστον λάβει δια της απουσίας Χαιρετίζω την παρουσία του εκπροσώπου της Λατινικής Προεδρίας και εκτιμώ αυτά που μας είπε. Απ' την άλλη μία όμως μιλάμε για μια χώρα με την οποία έχουμε στενές σχέσεις αλλά ο επικεφαλής της εκτορικής μας πολιτικής απουσιάζει. Το βέτο της Ρωσίας και της Κίνας είναι σημαντικό γιατί αυτές οι δύο χώρες ανέλαβαν την ευθύνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την προώθηση της διαμάχης. Αναλαμβάνω την ευθύνη για θανάτους εκατοντάδων πολιτών το καθεστώς αύξησε τις ε, προσπάθειες του, ε, του για θανατώσεις ε, μετά το βέτο αυτό. Οι Ρώσοι λένε ότι δεν θέλουν να αλλάξει το καθεστώς γιατί θεωρούν ότι το καθεστώς αυτό είναι νόμιμο. Εμείς όμως θεωρούμε ότι ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει 6.000 πολίτες δεν είναι πια νόμιμο, έχει υποσκάψει την νομιμότητά του. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες διπλωματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα βοηθήσει τους πολίτες που τη χρειάζονται, τους τραυματισμένους, τα θύματα επιθέσεων από κυβερνητικές δυνάμεις. Θα πρέπει να βοηθήσουμε εκείνους που δεν μπορούν να φτάσουν στο νοσοκομείο. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Ένωση τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Όσο πάει τόσο περισσότερο μας απαγοητεύουν οι εξελίξεις στην Συρία. Ακούσαμε εδώ στο σώμα να εκφράζονται ησυχίε από πολλές πλευρές. Βλέπουμε τα προβλήματα χιλιάδες πολιτών στη Συρία πεθαίνουν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από εκείνα που έχουμε κάνει, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα από τις διπλωματικές κυρώσεις, περιορισμένες οικονομικές κυρώσεις. Είναι μάλλον αληθές ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά έχουμε πρόσφατα α, παραδείγματα πως η διεθνής κοινότητα έδρασε όμοφωνα και διπλωματικά και στρατιωτικά με πάρα πολύ επιτυχές επιτέλεσμα. Ποιο είναι το νόημα μια τέτοια συζήτηση, ποιο είναι το νόημα ενό τέταρτου ε, ψηφίσματο για τη Συρία. Έχει νόημα γιατί πρέπει να εκφράσουμε την ελεγγύη μα με τη Συρία. Θα πρέπει να μάθει ο ηγέτης της Συρίας ότι τον παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε στενά το τι κάνει και φροντίζουμε θα φροντίσουμε μάλλον οι πράξεις του αυτές να μην μείνουν ατιμόρυτες. και θα ήθελα να καλέσω τους ε, επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευρύνουν τις κυρώσεις και τις πολιτικές και τις οικονομικές, να δώσουμε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που υποφέρουν, σε εκείνους που έχουν ανάγκη και επίσης να εκφράσουμε την αποφασιστικότητά μας στη σχέση μας με την ε, Ρωσία και την Κίνα για να τους πείσουμε να υιοθετήσουν το σχετικό ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη. Ο πρόεδρος κ. Ποτασίβιτς ε, έδωσε και το παράδειγμα της στήρησης του χρόνου. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Λένα Κολάρσικα-Μπομπίνσικα για δύο λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, υπήρξε πρόσφατα ένα κύμα ε, διαμαρτυρία στη Βόρεια Αφρική, η Αραβική Άνοιξη, αλλά τέτοια κλίμακα ε, σφαγής αθώου πληθυσμού όπως αυτό που βλέπουμε στη Συρία δεν το είχαμε ξαναδεί. Βλέπουμε και μαθαίνουμε να βασανίζονται μέχρι και παιδιά από το στρατό. Πρόκειται για άκρος ομές βιαιότητες. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει δράση ίσως ακόμη και χωρίς ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί μέχρι να ακολουθήσει η Κίνα και η Ρωσία ίσως να είναι αργά. Είδαμε τι έγινε με τον ΝΑΤΟ και τη Λιβύη. Δεν μιλάμε ε, μόνο για τον τερματισμό τη σύγκρουση, αλλά και για παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί ακόμη και μετά το πέρα αυτή τη κατάσταση. Δεν πρέπει να κολυσιεργήσουμε άλλο, γιατί αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει και στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να αποτρέψουμε λοιπόν τέτοια ε, γεγονότα στο μέλλον. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να σκεφτούν πώς μπορούν να συνεργαστούν και με τη Συριακή Αντιπολίτευση μετά ε, την ε, πτώση του Άσαντ. Θα πρέπει να ε, γίνουν σχέδια για μια σταθερή Συρία στο μέλλον. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με, την Αραβική, με τον Αραβικό Σύνδεσμο και να εξασφαλίσουμε την αποτροπή συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Δεν θέλουμε ένα δεύτερο Ιράκ. Θα πρέπει να βασιστούμε στο λαό της Συρίας που έχει το αίσθημα του δικαίου που θυσιάζει, βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει άλλους από τις ομότητες του καθεστώτος. Επεξεργαζόμαστε μια γραπτή δήλωση για να στηρίξουμε ακριβώς αυτά τα άτομα. Ας ελπίσουμε να τελειώσει σύντομα ο Συριακός εφιάλτης, αλλά πρέπει να υψώσουμε τον άστημά μας στο πλευρό αυτών που είναι υπέρ της δικαιοσύνης ε, στη Συρία συνάδελφο κύριο Γιώργ για δύο λεπτά. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη Συρία, η χρήση βίας, ε, είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να το καταδικάσουμε απερίφραστα και έχουμε ακούσει πολλά σήμερα. Εγώ όμως έχω το εξής ερώτημα στο μυαλό μου. Γιατί είναι τόσο ισχυρογνώμονες ε, οι κυβερνώντες. Γιατί ούτε μια υποχώρηση, ούτε ένα συμβιβασμό δεν κάνει ε, ο Άσαντ. Νομίζω ότι αυτό χρήζει εξήγηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια αξιολόγη απάντηση. Πρέπει ε, να ξέρουμε ότι δεν είναι ενωμένη, αλλά άκρως κατακαιρματισμένη η Συρία με πέντε ομάδες ε, να ζουν ε, δίπλα-δίπλα στην κοινωνία. Οι Αλεβίτες είχαν μονοπολί στην εξουσία μεταξύ των οποίων το σύστημα του οικογενειακό του Άσαντε. Οι Δρούζοι, οι Χριστιανοί και οι Σίτες είναι άλλες τρεις ομάδες που φτάνουν στο 30% του πληθυσμού. Η πλειοψηφία ε, στο κέντρο του ασαντικού κινήματος ε, είναι οι μουσουλμάνοι Σουνίτες ε, που έχουν στερηθεί όλα τα προνόμια. Τι φοβάται το, το καθεστώς, ότι θα υπάρξει σουνητική πλειοψηφία που θα πάρει την εξουσία και έτσι δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση ή άλλες ομάδες να περιληφθούν σε ένα ε, κράτος, σε μια χώρα την οποία θα κυβερνούν οι Σουνίτες. Βλέπουμε όμως να συνεχίζονται οι σκοτομοί. Ε, αν ε, δεν βλέπει καμία από τις ομάδες ωφέλη από την κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και βέβαια πάρα πολύ σημαντικό για το διακανονισμό αν θέλουμε να ισχύσει είναι να σεβαστούμε όλες τις μειονότητες. Τώρα δίνω το λόγο στην ε, συνάδελφο κυρία Μόνικα Λουίζα Μακοβέη για δύο λεπτά. Thank you, President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους άμαχοι αυτή τη στιγμή στην ε, ε, Συρία. Ε, και ξέρουμε ότι στην ε, Χόμς έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 300 άτομα από την αρχή του Φεβρουαρίου και πλέον έχουμε χάσει και την δυνατότητα μέτρησης των θυμάτων. Παιδιά συλλαμβάνονται και ε, βασανίζονται. Ε, είναι ε, ατρόμητος ο Άσαντ μπροστά στο λαό του και μπροστά στην διεθνή κοινή γνώμη. Επομένως θα πρέπει να, ε, να σταματήσει οποιαδήποτε προμήθεια ε, προς, ε, προς την χώρα αυτή. Θα πρέπει να αυξηθούν οι κυρώσεις προς όλα τα μέλη των οικογενειών που καταγράφονται ως σύμμαχοι του Άσαντ και οπωσδήποτε θα πρέπει να ανοίξουν λεωφόροι ανθρωπιστικές έτσι ώστε να προωθηθεί η βοήθεια προς την Συρία. Ε, και θα πρέπει να πιεστεί ο Άσαντ να φύγει και να υπάρξει καλή και ειρηνική μετάβαση προς τη δημοκρατία. Δίνω το λόγο στην κυρία Αντρικένε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι προφανές ότι το καθεστώς του Μπασάρ Ελάσαντ διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και θα πρέπει να σταματήσουν αυτά αμέσως. Θα πρέπει ε, τα Ηνωμένα Έθνη μέσω του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, να, τα, να σταματήσουν. Θα πρέπει να συνεργαστεί ε, και ακόμα και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έτσι ώστε αυτές οι ομότητες να μην μείνουν ατιμόρυτες. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ε, είχαμε ε, την ικτρή στάση της ε, Κίνας και της Ρωσίας που μέσω βέτο μπλοκάρισαν το ψήφισμα καταδίκησε της Συρίας. Εν τω μεταξύ σκοτώνονται οι άμαχοι εκεί. Ε, λόγω της στάσης των δύο αυτών χωρών, το ε, Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ε, δεν κατάφερε να καταδικάσει όπως έπρεπε το καθεστώς Άσαντ. Αναμφίβολα βλέπουμε ότι είναι στον επιθανάτιο ρόχο η κυβέρνηση Άσαντ. Επομένως θα πρέπει να στηρίξουμε τις διπλωματικές προσπάθειες της Βαρόνης Άστον. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Πάσκου. The Η γενική εικόνα της αραβικής ε, ανάπτυξης, ε, η, Συρία διχάζει το Ενωμένο το Συμβούλιο Ασφαλείας. Άλλοι στηρίζουν το ψήφισμα, άλλοι όχι. Εάν κάποιοι θέλουν ε, απλά να υπάρξει ξένη παρέμβαση, ε, υπάρχουν και άλλα κίνητρα που τα βλέπουμε να τα έχει η Ρωσία, η οποία είναι ένα στρατηγικό εταίρο, είναι μέσα στην εξίσωση στη Μέση Ανατολή, είναι επίσης και σημαντικός πελάτης για τις εξαγωγές ε, όπλων. Έχει πολύπλοκες σχέσεις και με το Ιράν. Η βέβαια η διεθνή κοινότητα στο μεγαλύτερο βαθμό, ε, στο μεγαλύτερο μέρος είναι κατά του καθεστώτο ε, του Άσαντ. Μην φτάσουμε στο σημείο που πλέον ε, θα έχουν αντραπεί όλες οι ισορροπίε. Χριστίνα Όγιουλαντ, για ένα λεπτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με την και κυρώσεων στη χώρα αυτή. Λυπούμε που η Ρωσία και η, Κίνα δεν ε, συνέβλεψαν για το ψήφισμα στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Θα πρέπει να δείξουμε άνευ ορών υποστηρίξη εκείνων που αντιτίθενται σε αυτό το καθεστώς. Στο περασμένο έτος είδαμε ότι ε, η βούληση των λαών μπορεί να αντιστρέψουν οποιοδήποτε καθεστώς οι συνάδελφοι προτείνουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα για το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να χρονοτριβούμε και να δώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της στρατηγικής που θέλουμε να ακολουθήσουμε προς τη Συρία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε στη Συρία ε, το, την φρίκη των όσων συμβαίνουν, αλλά διαφαίνεται παρόλα αυτά και η δυνατότητα να χυθεί ακόμα περισσότερο αίμα εάν διευρυνθεί ε, ο πόλεμος στην περιοχή. Ε, θα πρέπει να πιεστεί τουλάχιστον η Ρωσία ε, για να ε, σταματήσει την ε, στήριξη αυτή που έχει δώσει στον Μπασάρ Ελάσαντ λαμβάνοντας υπόψη και ότι στους δρόμους της Συρίας συνεχίζεται η αιματοσυχησία και λαμβάνοντας υπόψη τον βομβαρδισμό της Χόμς είναι απαράδεκτο να στηρίζεται η κυβέρνηση αυτή και βεβαίως αναρωτιόμαστε τι θα γίνει και στο μέλλον μέλλον. 2,5 ε, εκατομμύρια ε, χριστιανοί στην ε, Σύρια ε, βλέπουν ότι η θέση των χριστιανών δεν έχει γίνει πιο εύκολη στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στην Τινησία και ότι αυτή η Δημοκρατική Αυγή δεν, τους, δεν συμπεριλαμβάνει και τους χριστιανούς θα πρέπει να προστατευτούν οι μειονότητες και διεθνείς εγγυήσεις να δοθούν κατά αυτήν την έννοια. Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου, όσο πάει περισσότερο αυξάνονται οι ενδείξεις ότι η διένεξη στην Συρία θα γίνει αυτή η πυρκαγιά θρησκευτική βάσης που φοβούνται πολύ. Είχαν βοηθήσει στο Ιράκ, τώρα θα υπάρχει το ίδιο στην Συρία. Γιατί η κοινή θρησκεία ότι και οι Σουνίτες στην, ε, στα σύνορα του Δυτικού Ιράκ προσπαθούν να ε, δυναμώσουν τη θέση τους και έναντι της κυβέρνηση της Βαγδάτης. Σαν να μην ήταν αρκετά όλα αυτά, τώρα βλέπουμε ότι και η Αλκαΐδα θέλει να αναμειχθεί στην Σύρια. Κατά τη γνώμη μου, λόγω του ρωσικού βέτο, μία αποστολή και ανοφόρων δεν θα είχε πολλές δυνατότητες επιτυχίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να μην εμπλακεί περισσότερο σε αυτή την δίνη συγκρούσεων γιατί το μόνο που θα μπορέσει να καταφέρει είναι να καεί και η ίδια και να αποτύχει παραγωγών. Ε, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βίλη, εξ ονόματος Αντιπροέδρου της Επιτροπής και υπάτης εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. The floor is yours. Øh, Πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν πάρα πολύ ε, καλή αυτή η συζήτηση και ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη. Νομίζω ότι όλοι εδώ στην αίθουσα συμμερίζονται την ίδια ε, άποψη. Δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλο, δεν μπορούμε να αντέχουμε άλλο, να βλέπουμε ανθρώπους να βομβαρδίζονται, ε, να πυροβολούνται άτομα που διαδηλώνουν ειρηνικά, να μασανίζονται, να εξαφανίζονται, να πρέπει να εγκαταλείψουν τις πόλεις τους. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε ε, την καταδίκη και τον αποτροπιασμό μας απέναντι σε ένα καθεστώς που ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους εμείς στο Συμβούλιο έχουμε αξιοποιήσει όλες τις συναντήσεις μας ε, από τότε που θυμάμαι δηλαδή για να ε, συζητήσουμε το θέμα της Συρίας. Πάντα η Συρία ήταν στο, στην ημερήσια διάταξη και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πω ότι έχουμε στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική αυτή είναι αυτή η οποία μας ε, καθοδηγεί και θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί. Θέλουμε να βοηθήσουμε ε, από τις παρούσες συνθήκες όσο δυνατόν περισσότερο τον πληθυσμό της Συρίας. Πρώτη εντολή. Ε, πρέπει να σταματήσει η βία. Και αυτή είναι και η συμβουλή μας προς το καθεστώς. Μην πυροβολείτε το λαό σας, τους δικούς σας ανθρώπους. Ε, και άλλωστε αυτό το λέμε και σε οποιοδήποτε βήμα, διεθνές βήμα συζήτησης, ε, όπως τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα εκεί θα ψηφίσουν αύριο ένα ψήφισμα που κατά πάσα πιθανότητα θα καταδικάζει αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στη Συρία και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών γιατί ε, είναι σημαντικό και αυτό να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτό το είπαν και πολλοί ομιλητές. Ασκούμε επίσης κριτική στην ε, θέση της Κίνας και της Ρωσίας σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και απλά να παρακολουθούν αμέτωχοι τα τεκτενόμενα στη Συρία. Έχουν την υποχρέωση να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό. Το είπαν πολλοί ομιλητές αυτό. Θέλουμε να ε, θυμίσουμε το καθήκον αυτό στη Συρία και τη, στην Ρωσία και την Κίνα. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που το λέει και αυτό ε, προκαλεί εντύπωση. Το λέει η Τουρκία, το λέει και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Κινέζοι ε, σε ένα γύρο ε, στις ε, αραβικές χώρες έχουν ένα πρόβλημα για να εξηγήσουν την κατάσταση και για τη συμπεριφορά τους στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Τινησία, στην Τίνιδα, στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε μια συνάντηση εκεί και εκεί επίσης θα επαναλάβουμε τη θέση μας ότι πρέπει να σταματήσει η βία. Μόνο πολιτική λύση υπάρχει στην κρίση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Και θα κάνουμε ό,τι έχουμε πράξει σε οποιαδήποτε άλλο διεθνές βήμα συζήτησης. Αυτή είναι η δουλειά μας ως Υπουργείο Εξωτερικών και η δουλειά της κυρίας Άστον επίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δράσεις, γνωρίζω ότι αν υπομονείτε. Τέσσερις είναι οι πιθανοί τομείς δράσης. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτούς. Πρώτα απ' όλα, ο Αραβικό Σύνδεσμο, οι χώρε ε, οι αραβικέ πρότειναν να δημιουργηθεί μια ειρηνευτική δύναμη. Θέλουν υπό την αιγίδα όμω των ΗΠΑ να επιχειρήσει αυτή η δύναμη. Δεν ξέρουμε ακριβώ ε, πώ το σκέφτονται, θα μα τα διευκρινίσουν ε, στην τίνιδα αυτά. Δεύτερον, διεθνή διάδρομη, ανθρωπιστική διάδρομη. Δεν θα απέκλεια ε, τους αλλά πρέπει αυτό να το στηρίξει στεναρά η διεθνή κοινότητα. Γιατί πρέπει κανεί να πολεμήσει για να ανοίξει διαδρόμου. Γιατί και αυτό μιλάμε εδώ. Γίνεται πόλεμο. Γίνονται μάχε στη Συρία. Κάποιοι από του ομιλητέ επίση υπογράμμισαν τη σημασία τη αποτροπή ενό εμφυλίου πολέμου. Υπάρχει όμως αυτή η απειλή Ίσως λοιπόν το να μπουν περισσότερα όπλα δεν θα ήταν η βέλτιστη λύση, γιατί εκεί μπορεί να γίνει ανεξέλιγκτη πλέον η κατάσταση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η σημερινή συζήτηση επιβεβαιώνει την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνουν πιο αυστηρές οι κυρώσεις ε, και στις 27 ε, θα το ε, προωθήσουμε αυτό το μέτρο. Επίσης αυτές οι κυρώσεις ε, θα καλύψουν περισσότερα άτομα, ιδιώτες αλλά και ε, φορείς, οντότητες, εταιρείες. Δεν θα αποκλείσουμε κανέναν. Θα συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά με την ε, Συριακή Αντιπολίτευση και θα την καλέσουμε να ενωθεί, ώστε να μην είναι διχασμένη, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη Νέα Σύρια, να μην υπάρχουν διαιρέσεις και διχασμοί. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω. Ποια είναι η εναλλακτική λύση αντί του Άσαντ. Κάποιοι ανέφεραν ότι μπορεί μια εναλλακτική ε, να είναι ε, οι εξτρεμιστέ. Εγώ δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι οι Σύριοι θέλουν να ζήσουν όπως όλοι οι άλλοι. Θέλουν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Και εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Καμία χώρα δεν είναι καταδικασμένη να είναι δικτατορία ή να κυριαρχείται από ε, θρησκευτικούς εξτρεμιστές. Και η επιλογή τη χώρα στην οποία θα γίνει συνάντηση 24 στην Ισία, δηλαδή, νομίζω το επιβεβαιώνει αυτό, γιατί έχουμε δει εκεί αντίστοιχα πράγματα. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Θα διαβιβάσω ό,τι άκουσα στην κυρία Άστον, που φαντάζομαι το λάβει υπόψη και για το σχηματισμό, για τη διαμόρφωση ε, των επιχειρημάτων και τη θέση Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα έξι προτάσει ψηφίσματο για την περάτωση αυτή τη συζήτηση. κυρίω περιομένη τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 ώρα το μεσημέρι. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής